Bueno, si les Λοιπόν, να συνεχίσουμε, αν θέλετε. Και προχωρούμε. Αρχίζει η κανονική τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας με τα θέματα που έχετε στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 1. Ε, πρώτο, έγκριση ημερήσια διάταξη. Συμφωνείτε όλοι και όλες. Ωραία. Στο δεύτερο σημείο. Έγκριση των πρακτικών ε, των προηγουμένων συνεδριάσεων. Τα έχετε. Δεν ξέρω αν έχετε καμία έσταση, αλλιώς θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ωραία, εγκρίνονται. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι η συνεδρίαση των συντονιστών συμφώνησε για το ετήσιο πρόγραμμα ερευνών για το 2017, για τα εργαστήρια, για τις, τα ενημερωτικά σημειώματα και τις μελέτες. Το επόμενο θέμα ήταν της κυρίας Μαρινάκη που μόλις διεκπαιρεώσαμε για το 4 και πάμε στο 5 που είναι η συστάσεις προς το Συμβούλιο για την Επιτροπή του Καθεστώτος των Γυναικών. Οι, συγγητές, οι είναι δύο, η κυρία Λεγκρίπ και η κυρία Ρενά. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ρενά. Η κυρία Λεγκρίπ μαθαίνουμε ότι θα απουσιάσει σήμερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Είναι μέσα στην ίδια λογική με την ε, συζήτηση που μόλις κάναμε με τη Μάρα. Και πραγματικά ήταν μεγάλη μου χαρά να ακούσω την παρουσίαση της εκπροσώπου της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που ξεπερνά ακόμα και τις φιλοδοξίες των συστάσεων που είχαμε συντάξει για την έκθεσή μας. Χαίρομαι λοιπόν προκαταβολικά για τη συνεργασία που θα έχουμε τις ερχόμενες εβδομάδες μαζί της και στην όλη διαδικασία της συζήτησης για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προβάλλει κι άλλο τις δικές της προτεραιότητες για την 61η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ. ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτή τη έκθεση, υπενθυμίζουμε κάποιε προτεραιότητε. Προτεραιότητε τη Ένωση που υποστηρίζει και το Ευρωκοινοβούλιο γύρω από πέντε βασικά θέματα. Το ένα είναι η γενικότερη προσέγγιση για τα θέματα της ισότητας ανδρών γυναικών. Το θυμίζουμε απλώς γιατί ακόμη και αν αυτή η Γενική Αρχή έχει ενσωματωθεί στις συνθήκες, στις συμβάσεις και τη διεθνή νομοθεσία, δυστυχώς αποδεικνύεται ότι ακόμα και στην Ευρώπη η υλοποίηση αυτής της αρχής της ισότητας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ούτε γίνεται με τέλειο τρόπο. Καλό είναι λοιπόν να το θυμίζουμε εδώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο διεθνές προσκήνιο όπως στον ΟΗΕ. Ως προς τη γενική λοιπόν προσέγγιση στα επίπεδα της έκθεσης υπάρχει έτοιμα προς το Συμβούλιο να ε, αναλάβει δέσμευση για να προωθήσει κι άλλο την ατζέντα του Πεκίνου, να διευκολύνει την επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών, να καταπολεμήσει τη βία, να προβλέψει την οικουμενική πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλική και αναπαραγωγικής υγείας και για τα γενετικά δικαιώματα να τα θυμόμαστε, να τα θυμίζουμε όλα αυτά. Έπειτα υπάρχει η βελτίωση της ε, ανεξαρτητοποίησης των γυναικών από οικονομική σκοπιά και όχι διακριτική μεταχείριση στην πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. Θυμίζω αυτά που είχαμε πει για τις διαφοροποίησεις τις μισθολογικές και τις συνταξιωτικές όμως και ένα θέμα όπως η ισότιμη κατανομή των οικοκυρικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Κάτι που μας φέρνει και στο θέμα στην της πρόσβασης της γονικές άδειες και άδειες μητρότητας. Αλλά και στη διευκόλυνση των ε, πιστώσεων. Θα πρέπει να είναι ισότιμη η συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ε, λήψης αποφάσεων. Και αυτό συνδυάζεται με αυτό που έλεγα και προηγουμένως για τα φαινόμενα πολιτικής βίας. Είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Όχι απλώς γιατί εμείς οι ίδιες είμαστε πολιτικές γυναίκες και άνδρες, αλλά γιατί ε, περιορίζεται το ελεύθερο πεδίο για τους ανθρώπους που θέλουν να εκφράσουν ε, την ε, συμφωνία τους με την πράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Έπειτα να ευνοηθεί η πρόσβαση των γυναικών στη γη και την κατοχή γης στις περιοχές της υπαίθρου υπάρχουν εκεί γυναίκες ιδιαίτερα ευάλωτες να προωθηθεί η έγκριση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες, η πρόσβαση των ε, γυναικών προσφύγων στις θέσεις εργασίας και των εκτοπισμένων το ίδιο. Ένα φαινόμενο που δεν συζητείται πολύ στην Ευρώπη, γιατί ε, εδώ μιλάμε πολύ για τις πρόσφυγες, αλλά είναι μειονότητα σε σχέση με τις εκτοπισμένες γυναίκες. Είναι απλώς η κορυφή του, η παγόβουνου ε, σε σχέση με το συμβαίνει στις πέντε υπήρους. Θα πρέπει λοιπόν ε, ε κάποια μέρη να αναλάβουμε και εμεί στο Ευρωκοινοβούλιο να φροντίσουμε στη διαδικασία λήψη αποφάσεων οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΟΗΕ από την σχετική και αρμόδια επιτροπή να συνδυάζονται με αυτές τι αρχές που εκφράζουμε. Έτσι λοιπόν εμεί ω ευρωβουλευτέ έχουμε έναν ιδιαίτερο ρόλο εκπροσώπησης των ευρωπαϊκών λαών και θα πρέπει όλα αυτά να αντικατοπτρίζονται στη δουλειά της επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών, ώστε να δοθεί απαραίτητη προβολή και στο διεθνέ προσκήνιο, όπω έλεγα, στον ΟΗΕ και να δείξουμε ότι οι πολιτικές θέλουμε να χαράσονται και σε εκείνη την ε, περίπτωση. Αυτά, Πρόεδρε, σε σχέση με αυτή την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι βλεπόταν ολοκληρωθεί ω το τέλο τη χρονιά. Μπορούμε να παρατείνουμε λίγο την ε, προθέσμα για την υποβολή των πολιτιών και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και εγώ και η Κωνσταντ για τα όσα θα υποβληθούν, διότι κάθε μια και ο καθένα θέλουμε να συμβάλλουν. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρενά. Όπως λέτε λοιπόν και εσείς ενημερώνω ότι υπάρχει μια τροποποίηση σε ό,τι αφορά την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών από ε, ε, αυτή που ίσχυε 11 Ιανουαρίου πλέον 12 το μεσημέρι. Η νέα προθεσμία έρχεται ακόμα λίγο χρόνο παραπάνω. Και τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Κυρία Thank you. Thank you, um, Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τις δύο συνεισηγήτριες για την έκθεση αυτή. Ε, πολύ διεξοδική. Να θυμηθούμε κάποια σημεία που μας θύμισε και η Μαρία. Ε, η βία κατά των γυναικών και κυρίως η εμπλοκή του στην πολιτική. Ένα θέμα που δεν έχουμε συζητήσει ακόμα είναι η επιγραμμική βία. Ε, η κατάχρηση και η παρενόχληση των γυναικών ε, με πολλούς τρόπους στο ίντερνετ, στο Twitter, ε, με email. Υπήρξαν πολύ προβεβλημένες περιπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα θέματα αυτά. Και επειδή προέρχονται από αόρατες πηγές, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μορφές βίας, πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτές. Γιατί αν δεν το θίξουμε εμείς οι γυναίκες, κανείς άλλος δεν θα το κάνει. Ευχαριστούμε κυρία Χόνιμπολ, κυρία Μπεθέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω πολύ απλά να πω ότι στηρίζω ε, την πρόταση Χάνιμπολ 100%. Πάρα πολύ ευστοχή και πολύ σημαντική πρόταση. Δεν είναι περιστασιακό, δεν είναι του σειρμού, είναι κάτι που ήρθε για να μείνει ως ε, ε, κατάσταση και πραγματικά πρόκειται για καταπάτηση δικαιωμάτων και πρέπει να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνη, Πρόεδρος. Ναι. Ε, βλέπω ότι και άλλες ε, συγκατανεύουν ε, και συμφωνούν με την κυρία Χόνιμπολ και την κυρία Μπεθέρα. είναι κοινό το πρόβλημα και γι' αυτό θα καταρρεθούν σχετικές τροπολογίες. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος ή κάποια άλλη συνάδελφος το λόγο, που δεν θέλει. Σα είπα ποια είναι η προθεσμία κατά τροπολογιών, 11 Ιανουαρίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μα στι 25 Ιανουαρίου και το Φεβρουάριο στην Ολομέλεια. Αν συμφωνείτε. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης για τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση. Συντάκτης της έκθεσης είναι ο κύριος Πιμέντα Λόπες. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχηθώ σε όλους τους παριστάμενους Καλή χρονιά. Ελπίζω να ήταν ευχάριστη η περίοδο των διακοπών με την οικογένειά σας και ότι όλοι εκμεταλλευθήκαμε αυτή την ανάπαυλα για να αναπνεύσουμε. Δεν έχω πολλά να πω για το έγγραφο. Είναι δύσκολο σε 1500 χαρακτήρες να καλύψει κανείς ε, δύο-τρεις ιδέες και να τις αναπτύξει πλήρως γύρω από αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Προσπαθήσαμε λοιπόν στην, ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης που θα συζητηθεί να μετουσιώσουμε όλες αυτές τις βασικές ιδέες. Δύο-τρεις είναι οι βασικές ιδέες, ιδέες κλειδιά τις οποίες θα βασιστούμε για να προχωρήσει το σχέδιο γνωμοδότησης. Πρώτα απ' όλα καταπολέμηση των ανισοτήτων και της διακριτικής μεταχείρισης, αυτό που να συνδυαστεί με την καταπολέμηση της ένδυας ε, ως τρόπο ε, τρόπος καταπολέμησης των ανισοτήτων ακριβώς και της διακριτικής μεταχείρισης, που ε, ιδιαίτερα απαντώνται στον ε, κόσμο, στον χώρο της εργασίας. Επίσης, οι συνθήκες εργασίας και η καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας, και η προστασία της ε, και της πατρότητας, δηλαδή της ιδιότητας του γονέα. Ε, στοιχεία που δέχονται πίεση λόγω αυτής της, λόγω των ανισοτήτων. Δύσκολο σε τόσο σύντομο κείμενο να ε, εκφραστούν και άλλες τόσες ιδέες που θα ήταν πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται. Η ανάγκη να υπάρχουν λεπτομερή και ποσοτικά στοιχεία για τις μορφές διακριτικής μεταχείρισης από τη μια και από την άλλη για τους τρόπους να αντιμετωπιστεί και να αναχαιτιστεί η ε, διακριτική μεταχείριση. Μόλις ε, συζητήσαμε εδώ την έκθεση της κυρίας Λεγκρίπ για την ε, απόκληση στα συνταξιδοτικά. Σημαντικό θα ήταν και στη δική μας την γνωμοδότηση να αναφέρεται. Ο αντίκτυπος των εργασιακών συνθήκων και της επισφαλούς εργασίας ακριβώς στην τελική απόκληση και στις συντάξεις. Όμως θα θέλαμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ε, μητρότητα μέσα από τις δημόσιες, τις κρατικές πολιτικές που να εγγυώνται τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί ε, να ασκηθεί και αυτό το δικαίωμα. Σίγουρα θα είναι πολλές οι έννοιες που θα λείψουν από, την, ε, από το σχέδιο γνωμοδότησης εν τέλει και τα οποία ε, μπορούμε θεωρητικά να τα σκεφτούμε εύκολα, ε, πιστεύω ότι θα συνεισφέρουν όλοι οι σκιώδεις εισηγητές και όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, ώστε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς τους χαρακτήρες, τους τυπογραφικούς περιορισμούς. Είναι πολύ μικρή έκταση το κειμένο για να τα καλύψουμε όλα. Τελικά ελπίζω ότι θα παράξουμε μία γνωμοδότηση συνεκτική που θα περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της έκθεσης που θα θέλαμε να συντάξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιμέντα. Και τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις των συναδέλφων των μελών της Επιτροπής μας. Κυρία Αρένα. Απλώς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Αγιάλα Σέντερ, η οποία ψηφίζει αυτή τη στιγμή σε μια άλλη επιτροπή. Και δεν μπορεί να είναι δυστυχώ εδώ, ε, ως και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ε, δεν έχω και τι παρατηρήσεις της, να τι διαβάσω ζητώ συγγνώμη. Η κυρία Ζαμπόσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Στηρίζω τις προσπάθειες ε, του εισηγητή και συμφωνώ με την τοποθέτησή του. Πρέπει να βελτιωθεί η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Υπό αυτήν την έννοια ε, θεωρώ τις προτάσεις του ενδιαφέρουσες διότι μιλά για απόκληση στα μισθολογικά, στην διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, που παίρνουν διαφορετικούς μισθούς για ίση εργασία. Το γεγονός που επεσήμανε ο εισηγητής ότι πολύ συχνά οι γυναίκες είναι κατεξοχήν εκείνες που εκτός από τη δουλειά τους πρέπει να προσφέρουν και την φροντίδα των ανηλίκων είναι σαφής μορφή ε, διοικητικής μεταχείρισης στο επίπεδο της εργασίας. Οι γυναίκες που είναι και μητέρες αναζητούν τις ατυπικές συμβάσεις εργασίας για να βρουν κάποιο σημείο ισορροπίας μεταξύ του οικογενειακού και του επαγγελματικού τους βίου. Ε, να βρουν το χρόνο να αφοσιωθούν και στην οικογένειά τους. Ο εισηγητής αναφέρθηκε και σε αβεβαιότητες, σε ανασφάλειες. την ευελιξία που απαιτείται από τις γυναίκες. Η ευελιξία θα έπρεπε να προωθείται στην αγορά εργασίας αν πρόκειται για ελεύθερη επιλογή, για θελούσια επιλογή των γυναικών. Αν υποχρεούνται όμως να έχουν μια σύμβαση μη κλασικού, κλασικής μορφής οι γυναίκες από τον εργοδότη τους, εργοδότη τους, αυτό είναι τιμωρητικό. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη κατανομή του πλούτου, των πόρων όπως τους ονομάζει ο εισηγητής. Αυτό ίσως και περνά κάπως τα όρια του όσων θέλουμε να αναφέρουμε εδώ και το πεδίο εφαρμογής του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ίδιου και της ε, γνωμοδότησης. Πάντως, τα συμπεράσματα ο εισηγητής ζητά νέα νομοθετική πράξη από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα ε, το, της μητρότητας, πατρότητας και των γονεϊκών αδειών ζητάτε να αναλάβει πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υποβάλει νέα πρόταση. Ε, πρέπει να πω ότι κατεξοχήν η δική μου η ομάδα, η ομάδα των ε, χριστιανοδημοκρατών στην Ευρώπη, δεν θα ήθελε να υπάρξει ένα τέτοιο νομοθετικό ή μη νομοθετικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέτος. Και εγώ η ίδια πρέπει να πω ότι έχω ενδιασμού, έχω σοβαρού ενδιασμού ω προ την πρόταση αυτή του εισηγητού. Διότι από τη μια πιστεύω ότι θα ήταν επιζήμιο το Κοινοβούλιο να στραφεί αυτή τη στιγμή προς τα κράτη-μέλη ζητώντας ε, να προχωρήσουν σε έγκριση νέας νομοθεσίας. Οι δικές μας αρμοδιότητες στο νομοθετικό επίπεδο περιορίζονται από τις συνθήκες. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστούμε τα όρια που μας έχουν τεθεί. Ως προς την οδηγία για την άδεια μητρότητας, να επαναλάβω ότι η ελάχιστη διάρκεια των αδειών μητρότητας είναι ένα θέμα που έχει να κάνει πάνω απ' όλα με την υγεία της μητέρας και του νεογνού. Και είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής. Το να συνδυάζουμε όμως τις άδειες μητρότητας πατρότητα και τις γονικές άδειε και όλα να μπαίνουν στο ίδιο σακούλι. Αυτό δείξε τελικά και στην συνολική απόρριψη της πρότασης για τις άδειες μητρότητας από τα κράτη-μέλη. Εάν δεν αλλάξουμε εμείς τη στάση μας για το θέμα αυτό, θα, θα είμαστε συνυπεύθυνοι ε, για το γεγονός ότι η κατάσταση των γυναικών κατά την άδεια μετρότητας είναι αβέβαιη και έχει μείνει στο παρελθόν, σε αυτό που ίσχυε πριν από πέντε χρόνια. Και πάλι να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, συμβολή του, για τις διαφορετικές του προτάσεις. Και θα συμβάλλουμε με τις τροπολογίες μας στη βελτίωση της έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαπόσκα. Η κυρία Κούνεβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα δώσω συγχαρητήρια στον συνάδελφο Ζωάο για την δουλειά που έκανε για την νομοδότηση αυτή. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν, και στον συνάδελφο Σρικιώτη που συνέταξε την έκθεση για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόληση. Ένα σύντομο σχόλιο και από μένα, αν και δεν ανοίγω στου σκιώδε εισηγητέ. Έχω όμω ζήσει και πληρώσει ακριβά το τίμημα τη επισφαλού εργασία. Ξέρετε, οι επισφαλεί συνθήκε εργασία δεν είναι φαινόμενο σύγχρονο. Για τι γυναίκε οι συνθήκε εργασία ήταν πάντα επισφαλεί. Πληρωνόντουσαν λιγότερα όταν οι ήταν οι πρώτε που απολύονταν πιο επισφαλείς ήταν οι δουλειές εκείνες που θεωρούνταν πως ήταν επέκταση της γενικής τους φύσης, όπως για παράδειγμα οι θέσεις στον τομέα του καταρισμού ή της φροντίδας. Γυναίκες εργαζόμενες, αόρατες, προσωρινές, όχι μόνο για την εργοδοσία, αλλά και για την νομοθεσία που σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν τις προστάτευε στο παρελθόν και ακόμα και σήμερα δεν προστατεύει. Αυτό που σήμερα καλούμαστε να διαχειριστούμε είναι η αποτυχία της πολιτικής flex security ειδικά την Ελλάδα. Η λεγόμενη ευελιξία με ασφάλεια ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα εξαιτία των δανειακών συμβάσεων που κατόπιν συγκεκριμένων αποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρίθμισαν παντελώς τις εργατικές συνθήκες. Καλλιεργήθηκε λοιπόν στη χώρα μου και σε άλλες βεβαίως ευρωπαϊκές χώρες ένας φτηνός εργατικός πληθυσμός με περιορισμένες δυνατότητες αντίστασης εξαιτίας του φόβου της απόλυσης και την ανεργίας. Πώς να βάλουμε ένα στόπ στην επισφαλή εργασία λοιπόν. Προφανώς δεν γίνονται ταύματα από τη μια μέρα στην άλλη. Είμαι όμως αισιόδοξη πώς θα τα καταφέρουμε, γιατί στα δυόμιση χρόνια της θητείας μας έχουμε καταφέρει να εγκρίνουμε μια σειρά από κείμενα που είναι και σε καλή κατεύθυνση όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα η πλατφόρμα για την αντίοτη εργασία, η έκθεση για το οικιακό προσωπικό. Και τώρα, όπως θέλω να ελπίζω, διοτετήσουμε με μεγάλη πλειοψηφία την έκθεση και τι γνωμοδοτήσεις για την επισφαλή εργασία. Στα συνεχή κύματα εμφισβήτηση των αξίων της Ένωσης, το Κοινοβούλιο οφείλει να διασφαλίσει με κάθε τρόπο το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αν θέλουμε να μιλάμε ένα αληθινά κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κούνεβα. κυρία Μόντι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τη δουλειά του εισηγητή του κ. Πιμέντα και την στάση που έχει τηρήσει. Πιστεύω ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να προσθέσουμε σε αυτόν τον τομέα. ιδίω για την οδηγία για την άδεια για την επικυροποίησή τη και την θέση της σε ισχύ. Είναι ζωτική σημασία για μας. Ε, καθώς δουλεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς πρέπει να εκπροσωπήσουμε τους ανθρώπου. και να είμαστε βέβαιοι ότι προσφέρουμε βοήθεια σε αυτούς που τους ε, παγώνει ο κρύος, ε, ο παγωμένος αέρας αυτών των απάνθρωπων και ψυχρών πρακτικών της εργοδοσίας παντού. Υπάρχουν εντάσεις όμως και σε άλλους τομείς ε, και είναι και άλλες οι επιπτώσεις της επισφαλούς εργασίας όπως στην υγεία των εργαζομένων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον Υπάρχουν και οι συμβάσεις των μηδενικών ορών. Κάτι που κάνει πολύ δύσκολη την πρόσβαση στην φροντίδα των παιδιών, λόγου χάρη, την οργανωμένη φροντίδα των παιδιών. Θα καλωσορίσω λοιπόν το κειμενό σα και πραγματικά ευχαρίστω θα κάνω προσθήκε στην όλη εξέλιξη τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Γιάννα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να καλωσορίσω και να επενέσω τη δουλειά του εισηγητή. Ε, υπάρχουν κάποιες σκέψεις ε, που έχουμε να υποβάλουμε ε, στην έκθεση αυτή. Δεν είναι μόνο γλωσσικές οι παρατηρήσεις, είναι και θέματα αρχής. Στην ισπανική μετάφραση γίνεται λόγος για διάκριση με βάση το φύλλο που είναι η κλασική διατύπωση ε, και πώς να το πω, η πολιτική, η πολιτικός ορθή διατύπωση που χρησιμοποιούμε ε, σε τέτοιες περιπτώσεις για τη διαφορά και τη μεγαλύτερη επισφάλεια που αντιμετωπίζουν στη δουλειά οι γυναίκες. Αλλά και σε άλλες μεταφράσεις ε, αυτό αναφέρεται διαφορετικά. όχι διακρίσεις βάση το φύλλο, αλλά και διαφορά φύλλου. Ξέρω εγώ μπορεί να είναι κάποιο προβληματικό εδάφιο. Ε, δεν είναι γλωσσικό αυτό, είναι και θέμα ουσίας και αρχής. Συμφωνώ με την ανάγκη να επιμείνουμε σε κάποιους ε, ε, τύπους, κάποιες φόρμουλες που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη και πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες. Ιδιαίτερα στην οικιακή εργασία, θα κάνουμε και τροπολογίε σχετικά, ε, ε, στην βοήθεια στο σπίτι και στην οικιακή εργασία είναι δύσκολο να ρυθμίσεις με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο τα πράγματα. Διαφέρουν ε, οι πραγματικότητες από χώρα σε χώρα, αλλά υπάρχουν καλές πρακτικές που μπορεί κάποιο να υιοθετήσει, που έχουν αλλάξει. Μετά την εφαρμογή τους έχουν αποδειχθεί στην πράξη αποτελεσματικές. Πολύ ωραία λοιπόν εντοπίζει τα προβλήματα ο εισηγητής και θα πρέπει να τα τονίζουμε αυτά και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθεια. Εδώ στο Βέλγιο υπάρχει ένα είδος εργόσιμου που λέγεται titre service και είναι μια επιταγή με την οποία πληρώνονται εκεί βοηθοί. Θα μπορούσε αυτό να βρει μιμητές. Στην Ισπανία ε, υπήρχε ένας νόμος, τον άλλαξε το Λαϊκό Κόμμα, ε, επανήλθε η επισφάλεια. Πάντως βελτιώσει υπάρχουν και με βάση τις βέλτιστες ή τις καλές πρακτικές μπορούμε να το ε, καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο των επισφαλών μορφών εργασίας. Θα κάνουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ και πάλι τον ε, εισηγητή για την έκθεση, την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γουόρντ. Ε, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν ε, ιδέες που σχετίζονται και με την έκθεση που είχα συντάξει εγώ. για το πώ θα πετύχουμε του στόχου καταπολέμηση τη ένδυα με το μικρότερο δυνατό κόστο. Πήραμε μέρο σε πολλές με ενδιαφερομένους και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το βάρο τη λιτότητα το πληρώνουν, ε, το τίμημα τη λιτότητα το πληρώνουν οι γυναίκες κυρίω. Και αυτέ φέρουν το βάρο αυτό. Είτε δουλεύουν είτε όχι. Και αν δουλεύουν πληρώνουν και αν δεν δουλεύουν πάλι πληρώνουν το τίμημα. Νομίζω λοιπόν και πραγματικά θα ήθελα να κοιτάξετε λίγο την έκθεση και τη δουλειά που είχε γίνει προκαταβολικά για να συνταχθεί. Θα ήταν πολύ χρήσιμη, γιατί δινόταν μεγάλη έμφαση εκεί στη δυνατότητα να μπορεί κανείς ας πούμε, να καλύψει έξοδο έξοδα ενέργειας. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της έκθεσης. Οι γυναίκες πολλές φορές δηλαδή πρέπει να λάβουν αποφάσεις του αν θα θερμάνουν το σπίτι, αν θα μαγειρέψουν και θα έχουν ζεστό φαΐ στο τραπέζι. Κάτι άλλο ε, είναι και η διαφορά πρόσβασης ανδρών και γυναικών στην υγεία και στο σύστημα αυτό ή την ψυχολογική, την ψυχική υγεία. Εδώ ε, είναι πολλές οι γυναίκες που καταβάλουν διπλό κόπο για να καταλήξουν στο ίδιο ποσό χρημάτων ενώ ταυτόχρονα ανησυχούν για το αν θα πάρουν ποτέ σύνταξη και εφόσον έχουν τις ανάλογες, ε, τα ανάλογα ένσημα ή όχι. Αυτά λοιπόν έχουν μεγάλη σχέση με την υγεία και την ε, καλή κατάσταση των ε, ανθρώπων. Πρέπει ως φεμινίστριες, ως ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών τώρα να τα λάβουμε υπόψη μας και αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Γουόρντ. Και η κυρία Ρέτκε τώρα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και από τη δική μα πλευρά ευχαριστούμε τον συγγητή για την σύνταξη τη έκθεση. σω να ξεκινήσω με μια γενικότερη παρατήρηση. Έχω την αίσθηση ότι επειδή υπήρξαν προβλήματα με την αύξηση τη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα τη επισφαλού εργασία έχει λιγάκι επισκιαστεί. Έχω την αίσθηση ότι η ανεργία είναι τόσο μείζον θέμα που μα απασχολεί τώρα, που αρκούσε να πάει ο καθένα να δουλέψει όπου να είναι. Και αυτό έχει δημιουργήσει καταστάσει όπου στη δική μου τη χώρα λόγω Γερμανία όλη αυτή η συζήτηση για τι επισφαλεί θέσει εργασία δεν έχει έρθει στο επίκεντρο ε, όπω θα έπρεπε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό τώρα να γίνει. Γιατί οι γυναίκε όντω ακριβώ την επισφαλή εργασία κυρίω απασχολούνται, απειλούνται από τη φτώχεια, από τι ανισότητε και με πολύ συγκεκριμένε μορφέ αυτών των ε, φαινομένων. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω ένα-δυο στοιχεία τα οποία θα τα αναφέρουμε και σε σχετικέ τροπολογίε. Πρώτα απ' όλα, οι δημόσιε υπηρεσίε αναφέρατε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην ε, φύλαξη των παιδιών και τι σχετικέ υπηρεσίε. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα με τι δημόσιε υπηρεσίε που θα πρέπει να προσφέρουν εδώ τι κατάλληλε υποδομέ και υπηρεσίε. Πολλέ φορέ ακριβώ οι συνθήκε τη δημόσια υπηρεσία έχουν να κάνουν με γυναίκε που αυτέ εργάζονται σε αυτού του χώρου με ε, επισφαλείς συμβάσεις. Λόγου χάρη γυναίκες που ε, πάνε τα παιδιά τους ε, σε κέντρα φύλαξης όπου εργάζονται γυναίκες με επισφαλείς συνθήκες. Εκεί πρέπει να φροντίσουμε ε, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη ε, μπορεί να, πει, να, να συγκρίνουμε το, την αμοιβή ενός ηλεκτρολόγου με κάποια νηπιαγωγό π.χ. και να δούμε πόσο τεράστια είναι η απόκληση. Μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό έχουν ρόλο όσοι εργάζονται ακριβώς στον τομέα της φύλαξης και της φροντίδας των άλλων και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλειας. Θα πρέπει να υπάρχει για κοινωνική ασφάλιση που να καταπολεμάται όντως μέσω αυτής η φτώχεια. Έχουμε συζητήσει εδώ διαφορετικέ επιλογές, διαφορετικά συστήματα αλλά κυρίω πρέπει να τονίσουμε περαιτέρω στην έκθεση ότι οι επισφαλίστε τη εργασία συχνά είναι Κάτι που εντείνει και το μισθολογικό και συνταξιδοτικό χάσμα μακροπρόθεσμα. Εδώ λοιπόν η ένδυα, ιδίω για τις μεγαλύτερες ηλικίε γυναίκες, είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να το δούμε με μια πρωτοβουλία μας ξεχωριστή κάποια στιγμή. Αλλά πρέπει να αναφερθεί. Και το άλλο είναι ότι σε πολλά κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων και η Γερμανία έχουμε ακόμα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που κυρίως δεν αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως ε, πλήρως απασχολούμενες. Τις αντιμετωπίζουν ως ε, άτομα που ε, κάτι συνεισφέρουν στο βασικό εισόδημα της οικογένειας που είναι κυρίως του άντρα. Πρέπει λοιπόν εδώ αυτό να τονιστεί. Οι γυναίκε, θα πρέπει εξατομικευμένα να προστατεύονται στο σύστημα κοινωνική ασφάλεια, ιδίω εάν απασχολούνται σε επισφαλείς συνθήκε. Θα πρέπει λοιπόν να ενδυναμώσουμε αυτά τα σημεία τη έκθεσης με τι σχετικέ τροπολογίε που θα υποβάλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρένκε και για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό θα δώσω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Πιμέντα. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Δεν θα απαντήσω σε όλες τις ε, συνεισφορές. Ε, Βεβαίω και θα αναμένω για καώ τις γραπτέ σα τροπολογίε, ώστε να ξεκινήσει η όλη δουλειά. Υπάρχουν όντω περιορισμοί στην πρώτη εκδοχή της γνωμοδότησης και έπρεπε να επιλέξουμε κάποιε από τι πρώτε ιδέε που ευχαρίστω μπορούν να μεταβληθούν κιόλα στη συνέχεια. Υπάρχουν πτυχέ που και για ιδεολογικού ε, λόγου θα μα βρουν κάπω με διαφορετικέ απόψει. Δηλαδή ανισότητες προκαλούν και κοινωνικές ε, διαφορές και αποκλήσεις όπου ακριβώς ε, υπάρχει ε, αντιπαράθεση των ίδιων των γυναικών. Σίγουρα θα έχουμε και ιδεολογικές λοιπόν αποκλήσεις και δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε 100% σε όλα, όλοι μεταξύ μας. Όμως, Νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρο του κειμένου δεν, θα υπα... δεν θα υπάρχουν προβλήματα, διότι οι αρχέ τι οποίε προασπιζόμαστε είναι κοινέ για όλου. Ε, και υπό την ίδια λογική, νομίζω ότι με μεγάλη πλειοψηφία θα καταφέρουμε να διατυπώσουμε και να εκφράσουμε ένα κείμενο με ιδέε που όλου θα του βρουν λίγο πολύ σύμφωνου και θα μπορέσουν να το στηρίξουν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Πιμέντα. Σα ενημερώνω ότι για τις τροπολογίες έχουμε προθεσμία τις 12 Ιανουαρίου και ώρα 3 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας ε, στις 6 Φεβρουαρίου, στην απασχόληση ψηφοφορία ε, θα γίνει μια εβδομάδα μετά και τον Ιούνιο θα ψηφιστεί η έκθεση στο Λομέλια. Επόμενη έκθεση κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων. Η κυρία Κλέρ Μούντιν, η συγγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους οι οποίοι υπέβαλαν τις τροπολογίες του στην έκθεση αυτή. 245 συνολικά ήταν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν και τώρα επεξεργάζομαι συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες θα σας στείλω και απόψε γιατί ε, Έχουμε ήδη συζητήσει και θα έχουμε και μέσα στη βδομάδα και μια ακόμα συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές. Πολλές από τις τροπολογίες εστίασαν ε, στον όρο ισότητα των φύλων. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Κονδύλια για την ισότητα των φύλων» ούτως ή άλλως. Σίγουρα βέβαια με τους συναδέλφους θα επεξεργαστούμε την ορολογία αλλά νομίζω ότι φαίνεται λογικό να χρησιμοποιήσουμε την ίδια ορολογία, την ορολογία του τίτλου της έκθεσης και στο σώμα της έκθεσης. Θα εργαστώ όμως επικοδομητικά με τους συναδέλφους και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμβιβασμούς για όσο δυνατόν περισσότερες τροπολογίες. Πιστεύω και ελπίζω να το δουν αυτό οι συνάδελφοι όταν θα τους ε, στείλω αργότερα σήμερα τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες ε, που θα είναι η πρώτη φάση της περαιτέρω επεξεργασίας συμβιβασμών για μια μεγιστοποίηση της συνεργασίας τους με τις άλλες πολιτικές ομάδες και ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν στο διετών καλύτερο συμβιβασμό πάνω σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ κυρία Μούντι. Θα ήθελε κάποιο συνάδελφος, κύριε Κεσμπόφσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από μέρους της ε, Μπάρμπαρα Ματέρα, της συναδέλφου, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε άδεια μητρότητας, επομένως δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Η Ματέρα, την οποία εκπροσωπώ, θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για το έργο της και ελπίζει και η ίδια ε, σε μια επικοδομητική συνεργασία και στις προσεχείς ε, συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών με στόχο τελικά να υπάρξει ένα καλό αποτέλεσμα στον τομέα αυτό των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων και θα στηρίξει τις ε, τροπολογίες εκείνες ε, οι οποίες ε, ζητούν μια μελέτη αντικτύπου ώστε να υπάρχει πραγματικά ισότητα των φύλων και να δούμε πού θα χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, να δούμε πού έχουν αποδειχθεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και πού όχι αυτά τα κονδύλια. Υπάρχουν επικοδομητικοί επικοδομητικές προτάσεις. Δεν θεωρούμε ως έλκο ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με αρκετές, με πολλές από τις τροπολογίες, με μοναδικό πρόβλημα κάποιες τροπολογίες, όπως παραδείγματος χάρη αυτές, οι οποίες λένε μιλούν για τις διαφορετικές ε, ε των και γυναικών. Δεν υπάρχουν μελέτες που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι θεωρητικά κάπως τα πράγματα έτσι, αλλά δεν ε, ισχύει από όλους αριθμούς. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες που μιλούν για την ισότητα των φύλων. σε όλα τα νοικοκυριά, ε, υπάρχουν και σε, σε όλους του, μάλλον σε όλα τα κονδύλια του προπολογισμού, να είναι ένα θέμα δηλαδή που θα διατρέχει όλο τον προπολογισμό, αλλά νομίζουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Ε, υπάρχουν και κάποια ζητήματα, όπως πολιτική αλληλείας, συμφωνίες με τρίτες χώρες κτλ. Αλλού ζητείτε εξωτερικοί εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία κατάρτιση του προπολογισμού. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δυνατόν και δεν νομίζω να ικανοποιηθούν και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Προπολισμών. Υπάρχουν διαφορετικά όργανα που εκπροσωπούνται τα κρατημέλη. Δημοκρατία, διαφάνεια και ευρύτατη συμμετοχή είναι ε, σίγουρα αρχές οι οποίες υποστηρίζονται αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Νομίζω ότι εδώ όλοι αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των γυναικών. Αλλά τώρα να πούμε ότι οι φυσικές καταστροφές πλήττουν περισσότερο τις νέες από τους άνδρες, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, πηγαίνει λίγο μακριά. Καλό θα ήταν ε, οι συνάδελφοί μας να μπορούν να υποστηρίξουν ε, πιστικότερα τέτοιου επιχειρήματα. Αυτά σε ό,τι αφορά και κάποιε τη επιτροπή τη ομάδα των Πρασίνων. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Σαμπόρσκα. Ε, κυρία Τροσίνσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα σας μιλήσω για τις δικές μου τροπολογίες ε, που απανούν στις αρχές και τις αξίες μου που έχω ταχθεί να υπηρετώ και στο Κοινοβούλιο και στην ομάδα μου. Η συγκήτρια μίλησε προηγουμένως για την έννοια του φίλου, την οποία εγώ απορρίπτω, απορρίπτω κατηγορηματικά. Το gender στα αγγλικά σημαίνει φίλο, το genre στα γαλλικά σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι προϊόν ιδεολογίας που λέει ότι ο άνθρωπος όταν γεννιέται δεν είναι ε, αγόρι ή κορίτσι, αλλά είναι κάτι που αυτοπροσδιορίζεται με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, της επιθυμίες και τις ορμές του οι άνδρες και οι γυναίκε έχουν τα ίδια δικαιώματα και τι δουλειά έχει εδώ ε, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ε, ταυτότητα. Θα επανέλθω λοιπόν για να σας πω ότι αποκλείεται η συζήτηση για την ισότητα ανδρών και γυναικών να είναι μια πρόφαση ε, και ένα προπέτασμα ε, καπνού για να χρηματοδοτείτε την καταστροφική μεταναστευτική σας πολιτική. Θα πρέπει να προστατεύουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια στην Ένωση βεβαίως. Ε, δεν θα πρέπει να περιφρονούμε ή να παραγνωρίζουμε τα δεινά που υφίστανται οι μετανάστριες, αλλά πρώτα να ασχοληθούμε με τις δικές μας γυναίκες ε, και μετά ε, με τα υπόλοιπα. Αυτές είναι τροπολογίες 187, 197 και 201. Θα τα ξανασυζητήσουμε στους σκιώδεις εισηγητές για τις συμβαστικές τροπολογίες. Και όπως γνωρίζετε όλες οι χώρες μας μαστίζονται από βαθιά οικονομική κρίση από το 2008. Θα πρέπει να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις για να εφαρμόζονται σωστά. Έτσι, τα κονδύλια που δίνονται ε, για την ισότητα των φύλων είναι πάρα πολλά μέχρι και επικίνδυνα. Τα χρήματα των φορολογημένων θα πρέπει να είναι στην υπηρεσία των φορολογημένων και όχι να ε, τα διασπαθίζουμε σε προγράμματα που είναι ποτισμένα ε, από ιδεολογίες. Η κυρία Χάνιβολ έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λίγο να επανέλθω στον ορισμό της λέξης gender, φίλο. Χρόνια ολόκληρα είμαι εδώ μέλος και τον βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Αυτό το θέμα είναι γλωσσικό. Ε, στα αγγλικά ε, γίνεται διαφορετική διάκριση. Άλλο είναι το σεξ και άλλο είναι το gender. Ε, και δεν χωράει καμιά παρεξήγηση το ίδιο πράγμα λένε και τα δύο. Ε, δεν ξέρω τι ισχύει σε άλλες γλώσσες. Σε τέτοιες εκθέσεις ε, όταν είναι ο εισηγητής ή η εισηγήτρια αγγλόφωνη έχουμε πρόβλημα με τις μεταφράσεις. Αυτό είναι η αγγλική λέξη gender, το φύλλο. Ε, πάντα είναι θέμα σύμβασης ότι, ότι κάνουμε τις εκθέσεις μας στη μετρική γλώσσα του καθενός. Θα παρακαλούσα να διατηρηθεί αυτός ο τίτλος ε, και αν βοηθάει να τον αφήσουμε παντού στα αγγλικά τον τίτλο, αν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά στις άλλες γλώσσες. Ελπίζω κάπως αυτό να διευκολύνει. Γιατί είναι κρίμα πραγματικά ένα, για μια τέτοια γλωσσική υπόθεση να την πληρώσει έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Χάνεβον, Η ε, κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για να είμαι ειλικρινή, δεν είμαι εγώ σκιώδη συζητητρία, αλλά η κυρία Τζαμπόρσκα αναφέρθηκε σε εμά, στην ομάδα μα και τις τροπολογίες που καταθέσαμε. Θα ήθελα σύντομα να απαντήσω και με χαρά να σας δώσω και περαιτέρω ε, βιβλιογραφία. Γιατί το φύλλο έχει γίνει πλέον μια κατηγορία για αναλύσεις και ίσως εδώ οφείλεται και η παρεξήγηση που παρατηρούμε χρησιμοποιούμε διάφορες κατηγορίες για να καταγράψουμε την ε, πραγματικότητα που ζούμε και ο προπολογισμό με βάση το φύλλο μας δείχνει ποια κονδύλια χρησιμοποιούνται περισσότερο για τους άνδρες ή για τις γυναίκες. Εμείς τι θέλουμε με τις τροπολογίες μας, να το διευκρινίσουμε και να πούμε μα δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, ίση κατανομή ε, των κοινοτικών κονδυλίων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και σε σχέση με αυτά που είπατε για την αλληλευτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ συχνά δίνονται κονδύλια σε αλληλείς άνδρες και γυναίκες. Να το αναλύσουμε, να δούμε αυτό πώς επηρεάζει διαφορετικά τις αλληλευτικές κοινότητες. Υπάρχουν κοινότητες που εξαρτώνται πάρα πολύ ε, από την αλληλεία. Αναφερθήκατε σε θεομηνίες, ε, πλημμύρες, σεισμούς. Συχνά οι γυναίκες αναλαμβάνουν την ευθύνη των ηλικιωμένων, των παιδιών που τα φροντίζουν και όταν πλημμυρίσει ο τόπος και χάσουν τα σπίτια τους, οι γυναίκες έχουν ψηλότερο ε, βάρος, μεγαλύτερο να σηκώσουν στους ώμους τους όταν φροντίζουν ηλικιωμένους και παιδιά. Εξού και η κατανομή των πόρων. Αυτό θέλαμε να μετρηθεί, αυτό θέλαμε να αναφερθεί. Υπάρχουν πολύ καλές μελέτες γι' αυτό. Αν θέλετε να σας τη στείλω για να διευκρινίσουμε γιατί έχει σημασία αυτό. Και ένα τελευταίο, δεν ξέρω αν είναι ιδεολογική συζήτηση που έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι αν θέλουμε πραγματικά να γίνει πραγματικότητα αυτό που λένε όχι μόνο οι συνθήκες, αλλά και άλλη ε, νομοθεσία για την ισότητα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η κατηγορία του φίλου. Και θέλω να ενθαρρύνω την εισηγήτρια να το χρησιμοποιήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, και ως όρος για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, να βελτιώσουμε την πραγματικότητα και να γίνουν οι πολιτικές έτσι ώστε η κοινωνία μας να είναι καλύτερη. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε και τι σημαίνει και το transgender και όλα αυτά. Ε, θα πρέπει ο ε, όρος gender να μην είναι ταμπού, να το χρησιμοποιούμε και να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε. Ευχαριστώ. Κυρία Ρένα. Euh, δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδεολογική ε, συζήτηση, ε, αλλά λένε κάποιοι ότι υπάρχουν καταστροφικές ιδεολογίες. Αυτό δεν μπορούμε να δεχθούμε. Και ότι αυτές είναι αυτές που μπορεί να καθορίζουν κάποια πράγματα. Όταν βάζουμε σε αντιπαράθεση τα δικαιώματα ορισμένων ανθρώπων, ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαίων, και τα αντιπαραβάλλουμε ανθρώπινα δικαιώματα άλλων, αυτό είναι καταστροφικό και καταστρέφει και τη συμβίωση. Οι γυναίκες λοιπόν σήμερα, οι οποίες βιώνουν επισφαλείς ε, συνθήκες ε, και διακριτική μεταχείριση παντού όπου βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και είτε είναι ε, από την Ευρώπη είτε από τρίτες χώρες, αυτές τις γης θα πρέπει να τις προστατεύσουμε. Δεν λοιπόν αντιτίθεμε από δημοσιονομικής πλευράς ή από πλευράς επιβολής μέτρων στο να μιλάμε για γυναίκες, είτε είναι Ευρωπαίες είτε δεν είναι Ευρωπαίες, μιλάμε για δικαιώματα και ανθρώπινα δικαιώματα αυτό πρέπει να το θυμίζουμε και είμαι πεπισμένη ότι πολλές Ευρωπαίες ε, είναι έτοιμες να το ακούσουν αυτό γιατί δεν θέλει κανείς να πεθαίνουν γυναίκες περιμένοντας ε, να υποστηριχθούν άλλες γυναίκες. Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο, και τις Ευρωπαίες και τις άλλες γυναίκες να τις υποστηρίξουμε ταυτόχρονα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πούμε διότι διαφορετικά αυτές οι καταστροφικές ιδεολογίες ε, θα δικαιωθούν και όχι οι άλλες, οι επικοδομητικές ιδεολογίες και νομίζω ότι εμείς στην πλειοψηφία μας ε, είμαστε υπέρ των θετικών πτυχών και όχι των αρνητικών πτυχών. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε τη συζήτηση με τη δευτερολογία της ηγήτριας κυρίας Κλέρ Μούντι. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω βέβαια για τα σχόλια του συναδέλφου σε σχέση και με τις ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι σε κάποιου τομεί ε, ίσως υπήρξαν κάποια μεταφραστικά προβλήματα σε σχέση παραδείγματο χάρη με το θέμα τη κυρία Ματέρα. Σε ό,τι αφορά τώρα το gender equality, ισότητα φίλων αν είναι ευρύτερο το θέμα ή καθαρά γλωσσικό, ε, υπάρχει ένα είδος, ε, μάλλον υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα που, είναι ότι αυτή η καθαρα γλωσσικο υπαρχει ενα μαλλον υπαρχει ενα πολυ χρησιμοποιείται στον τίτλο της έκθεσης και συνεχίζω να τη χρησιμοποιώ και στην έκθεση. Έτσι θεωρώ ότι είναι το σωστό. Και τον τίτλο τον συμφώνησε προηγουμένως η Επιτροπή. Δεν προσωπική επιλογή λοιπόν ο τέλος της έκθεσης. Ορισμένα από τα σχόλια, αρκετά από αυτά μάλλον, τα καλωσορίζω και σε κάποιες συμβασικές τροπολογίες τα έχω συμπεριλάβει. Συμφωνώ ότι εδώ μιλάμε για τη χρήση των φυστάμενων κονδυλίων και ιδίω ότι αφορά τι δαπάνε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Υπερπολογισμού. Παραδείγματο χάρη, όταν βλέπουμε το θέμα των προσφύγων, βλέπουμε τα κονδύλια που δαπανούνται ε, και είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να υποστηρίσονται οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο σε ομάδες αυτές κινδύνου. Όπως είπα λοιπόν και πριν, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλια ε, που διατύπωσαν και προσβλέπω στην συνέχιση της συνεργασίας μας με στόχο να μπορεί ε, να στηρίξει την τελική έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αμούντι. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης που είναι η αποστολή στην Ελλάδα. Το Νοέμβριο του 2016 επισκέφθηκε αντιπροσωπή της Επιτροπής μας στην Ελλάδα. Έχετε τα ε, σχετικά έγγραφα στο φάκελό σας συγκεκριμένα την έκθεση την αντιπροσωπείας. Βλέπετε ποια ήταν τα θέματα της μερικιάς διάταξης και κάποια συμπέρασματα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος το λόγο, αλλά μπορούμε να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση. Πρόκειται για απλή ανταλλαγή απόψε και όπως σας είπα έχετε και την έκθεση στο φακελό σας. Είναι σαφή τα πράγματα. Αν δεν έχετε κάτι να πείτε να περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι τα διάφορα. Αν δεν υπάρχουν διάφορα, δεν υπάρχει κάτι που θα θέλετε να επισημάνετε υπό τα διάφορα, περνάω στο επόμενο σημείο της που είναι η διεξαγωγή της επόμενης συνεδρίας της Επιτροπής μας, 25 Ιανουαρίου η ημερομηνία διεξαγωγής, 9 το πρωί. Και είναι και η συνεδρία σε σώμα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μας για σήμερα. Παναλαμβάνω τις ευχές μου προς όλους και όλες. Ελπίζω να είναι μια αποδοτική χρονιά για όλες και όλους, σε όλου τους τομείς. Και να συνεχίσουμε και εμείς ε, ε, και να φέρουμε σε αίσιο πέρα στι εργασίες μας. Σα ευχαριστώ και τα λέμε στην επόμενη συνεδρίαση.